Colleagues, please be seated. We still have two points of merit of this afternoon's agenda. Ε, καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι, απομένουν δύο σημεία στη σημερινή ημερήσια διάταξη, οπότε χωρίς άλλη καθυστερήση ας συνεχίσουμε. Το θέμα του επόμενου σημείου είναι στρατιωτική συνεργασία με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω στη συνεδρίαση μας, μας ε, τους τέσσερις, ε, τα τέσσερα μέλη του πάνελ, ε, τα τέσσερα εξέχοντα μέλη του πάνελ. Στα αριστερά μου ο, ο στρατηγός Αντρέι Φαλκόφσκι, στρατιωτικός εκπρόσωπος της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ. Έχουμε τον συνταγματάρχη Σερχή Ρέτσιτς, σύμβουλο σε θέματα άμυνας ε, στην αποστολή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έχουμε τον ε, συνταγματάρχη Γκίδης Καρδέλης, ε, αναπληρωτής εκπρόσωπο, στρατηγικός ε, εκπρόσωπος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ε, συνταγματάρχη Έρικ Χρέος. Ζητάει συγγνώμη Πρόεδρος επειδή δυσκολεύεται να προφέρει τα ονόματα. Αναπληρωτή εκπρόσωπο της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή, στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προηγηθεί μια μεγάλη μέρα διαβουλεύσεων με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς άλλη λοιπόν καθυστέρηση θα δώσω το λόγο με την ίδια σειρά με την οποία παρουσίασα τα διακεκριμένα μέλη του πάνελ. Ο στρατηγός Αντρέα Φαλκόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για αυτή την πρόσκληση. Να σας διορθώσω, δεν είμαι μόνο εκπρόσωπος ε, στο ΝΑΤΟ, αλλά και στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους δύο λοιπόν. Με την άδεια σας θα ήθελα να ξεκινήσω με, μια, ε, ε, με την παρουσίασή μου. Είναι 23 οι διαφάνειες, ορισμένες θα αφιερώσω μόνο ένα λεπτό ένα δευτερόλεπτο ώστε να μπορέσω να ε, τηρήσω το χρόνο των 8 λεπτών που θα χρειαστώ για να σας αναλύσω το ζήτημα. Ακούγοντα την παρουσίασή σας μάλιστα, ε, θυμήθηκα τη δική μου θέση στο Υπουργείο Άμυνας κάποια εποχή όπου ήμουν αρμόδιος για τον αμυντικό προπολογισμό της Πολωνίας. Ε, μια δύσκολη δουλειά, με έντονες συζητήσει τότε εκείνο τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της παρουσίασής μου Να σας δώσω δύο παραδείγματα της πρακτικής συνεργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο της παρουσίασης μου θα σας μιλήσω για τις μάχισμες ε, ε, Β' της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο θέμα θα είναι το τάγμα Λιθουανίας, Πολωνίας και Ουκρανίας ε, με αλφαβητική σειρά. Ας ξεκινήσω από τα βασικά. Εδώ βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα με τα βασικά. Οι μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα προέκυψε, γεννήθηκε το 2006 όταν, όπου προσδιορίστηκε η έννοια των μάχημων μονάδων και θα έχουμε εκδιπλωθεί πλήρως, ε, εκδιπλωθήκαμε ε, πλήρως το 2017. Έχουμε λοιπόν 10 χρόνια εμπειρίας. Ε, θα έχει αυτή τη μορφή λοιπόν, σύμφωνα με την αρχαιοκό προσδορισμό, 1500 ε, άτομα προσωπικού, ανάλογα με τις ε, απαιτήσει, ε, ανάλογα με την απειλή από που προερχόταν, τις απαιτήσει, ποιο σκοπό θα επιτελούσε. Κλασική λοιπόν δομή από που περιλαμβάνει υποστήριξη και υποστήριξη υπηρεσιών μάχης με όλες τις υπηρεσίες όπως αεροπορικές, διοικητική μέρημνα, θαλάσσιες ε, και τα λοιπά, ανάλογα με την περίπτωση. The European Union should be... Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να, μπορέσει, να μπορεί να λάβει απόφαση για την ανάπτυξη των μάχημων μονάδων εντός ε, πενθυμέρου. Δηλαδή ενεργοποιείται ε, η έννοια της διαχείρισης κρίσεων και σε αυτή την περίπτωση οι μονάδες πρέπει να είναι έτοιμες για επιχειρήσεις εντός του δεκαημέρου το οποίο είναι πολύ γρήγορο. Έχει προσαρμοστεί για την ελάχιστη στρατιωτική ε, αποτελεσματικότητα και για την αρχική φάση των 30 ημερών, 30 ημέρες διατήρηση. Ε, ό,τι χρειάζεται από τρόφιμα, από μέσα, από υπηρεσίες ε, αρκούν για 30 μέρες με δυνατότητα επέκτασης σε επιπλέον 120 μέρες σε περίπτωση ανεφοδιασμού. Ε, αρκετά λοιπόν ευέλικτη δύναμη θα έλεγα. Τώρα για λόγους προγραμματισμού βάσει ε, αυτό Ανάπτυξη αυτών των μαχημών μονάδων είναι 6.000 χιλιόμετρα από τι Βρυξέλλε ε, σε τέτοια ακτίνα. Φυσικά μπορούν να αναπτυχθούν οπουδήποτε, αλλά πρέπει ε, να πληρούνται ορισμένοι όροι. Τώρα, περιορισμοί και προκλήσει. Όπω ανέφερα πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα ε, έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2007, αμέσω αμέσως μετά από τον προσδιορισμό της Ολυσένειας και δημιουργήσαμε δύο ε, μαχημές μονάδες ε, εντός ενός εξαμήνου. Ε, πρώτη, η Γαλλία και το Βέλγιο έφτιαξαν μια μάχημη μονάδα το πρώτο εξάμεινο του 2004 ως βασικό έθνος ως έθνος πλαίσιο και μετά η Γερμανία ως έθνος πλαίσιο μαζί με τη Γερμανία και τη Φιλανδία δημιούργησαν δεύτερη μονάδα το ίδιο έτος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ, επειδή έχουμε μόνο ένα σύνολο δυνάμεων για όλα τα κράτη, αυτό που είναι ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι οι μαχημένες μονάδες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ επιχειρησιακά ε, σε επιχειρήσεις ε, των οποίων ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, έλλειψη πολιτικής βούλησης και πιθανώς και κάποιες απαιτήσει πόρων. Διότι όταν συζητάμε για προετοιμασία και περίοδο αναμονής, τα κράτη που παρέχουν τις δυνάμεις ε, Ε, πληρώνουν και το κόστος. Οπότε ε, για τη χρήση όμως τα πράγματα είναι κάτι, γίνονται διαφορετικά. My country. Η χώρα μου λοιπόν υπήρξε ε, κράτος πλαίσιο τρεις φορές Ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή μας στις μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 ως ε, κράτος πλαίσιο για τη Γερμανία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. Μετά το 2013 στο δεύτερο εξαμεινό Πολωνία, Γερμανία και Γαλλία ε, και τέλος πριν λίγο καιρό με το ε, μάχημη μονάδα ε, με τις τέσσερις χώρες του Βίσσεγκραντ. Πώς πήγαν τα πράγματα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το μέλλον. Όπως βλέπετε, έχουμε τον ίδιο σχηματισμό Βίσεγκρατ. Ε, συγγνώμη, κάποιος είπε κάτι. Ε, για το 2019 λοιπόν, το δεύτερο εξάμεινο έχουμε τον ίδιο σχηματισμό. Αλλά όπως βλέπετε από αυτόν εδώ τον πίνακα, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Έχουμε κενά ε, για το δεύτερο εξάμεινο του 2017 και για το ε, δεύτερο εξάμεινο του 2018. Τα κράτη δηλαδή δεν δείχνουν ιδιαίτερη βούληση να συμμετέχουν και να συμβάλλουν. Αν αλλίοντας αυτό το πίνακα ε, ουσιαστικά ε, βλέπουμε διαρκώς τα ίδια κράτη σε διαφορετικούς σχηματισμούς. Οπότε αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώ ε, ε, καταμερισμό του φόρτου. Ποια είναι η τελευταία μα εμπειρία την τελευταία φορά. Ε, πρώτα απ' όλα για πρώτη φορά είχαμε και ένα τρίτο μέρο, δηλαδή την Ουκρανία, που υπήρξε αρκετά γενναιοδορή ώστε να συμμετέχει στην ομάδα των τεσσάρων του Βίσεγκραντ. Που επισήμανε την ε, περιφερειακή διάσταση και εστίαση αυτή τη ομάδα. Τώρα η σύνθεση και οι δυσκολίες. Σύμφωνα με τους ορισμούς, με την αρχικό σχεδιασμό, προετοιμάζουμε τις ε, δυνάμεις μας ε, για τα καθήκοντα που αναφέρονται εδώ. Ε, αναγκαστικός διαχωρισμός μαχόμενων μερών, πρόληψη σειράξεων, επιχειρήσεις εκένωση, ανθρωπιστική βοήθεια, σταθεροποίηση, ανοικοδόμηση και στρατιωτικές συμβουλές. Αυτές είναι οι κλασικές ε, αρμοδιότητες ε, μάχημων μονάδων και είναι προετοιμασμένες οι μονάδες μας για την πλήρωση αυτών των καθηκόντων. Αυτό που δεν είχαμε ήταν τα, HQ, τα επιχειρησιακά, το επιχειρησιακό αρχηγείο. Κανονικά έχουμε στην Ευρώπη πέντε τέτοια πιστοποιημένα το Μαν Βαλεριάν στη Γαλλία, το Πόστονταμ στη Γερμανία, ε, το Λαρίσα στη Ρώμη, ε, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και τη στιγμή που φτιάχναμε όμως εμείς τη με μονάδα δεν μας ήταν διαθέσιμα. Χρειάστηκε λοιπόν να καταβάλουμε ποσά και στην Κρακοβία αναγκαστικά φτιάξαμε τα δικά μας το δικό μας επιχειρησιακό αρχηγείο το οποίο μας κόστησε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν χάθηκαν τα χρήματα γιατί το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον και για τους επόμενους ε, σχηματισμούς ε, αλλά ήταν κάτι που απέτυσε πολλά ειδικότερα σε θέματα υποδομής και υψηλής τεχνολογίας που θέλαμε να έχουμε. Σύνθεση τώρα. Η χώρα πλαίσιο παρέχει όλες τις δυνατότητες που δεν μπορούν να παρέχουν οι υπόλοιπες. Ε, πήραμε λοιπόν το 50% του βάρους από τις άλλες χώρες και χρησιμοποιήσαμε από τα άλλα κράτη, Ουγγαρία, Τσεχική, ε, Δημοκρατία, Σλοβακία και Ουκρανία, τις δυνατότητες που μπορούσαν να παρέχουν. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, ήταν αρμόδια για τις στρατηγικές μεταφορές. Πολύ, ε, στο πλαίσιο του ΑΝ 124 σχεδόν 4.000 ε, άτομα προσωπικού, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν. Και έγιναν και πολλά, γιατί δεν αρκούσε να πούμε ότι από τα ημερομηνία αρχίζουμε να ε, παίζουμε το ρόλο της μαχημής μονάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο χρόνια για την προετοιμασία διαφορές ασκήσεις σε εθνικό διεθνές επίπεδο, ασκήσεις πιστοποίησης τέλος και περίοδος αναμονής. Όλα αυτά είχαν σοβαρές απαιτήσει. Τώρα, τι ε, διδάγματα αποκομίσαμε από όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, μας δόθηκε η ευκαιρία σε περιφερειακό επίπεδο να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας όσον αφορά την εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και παντού. Δεύτερον, να προωθεί την περιφερειακή συνεργασία καθώς και την ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τρίτον, βελτιώνει, ενισχύει το στρατιωτικό συντονισμό με τέρους και η Ουκρανία εδώ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν μια πιο τυποποιημένη έννοια της μαχημής μονάδας διότι έχουμε 20 ετή εμπειρία και δηλαδή και εκεί 20 μαχημές μονάδες ήδη έχουν κάνει ασκήσεις οπότε έχουμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον. Τώρα όσον αφορά το κόστος ε, την κατανομή του κόστους του φόρτου. Μιλάμε τώρα για καταμερισμό του φόρτου, όχι του κόστους, του φόρτου. Και φυσικά θα θέλαμε να συμμετέχουν περισσότερες χώρες ε, στις ε, μάχημες μονάδες, εννοείται, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε τις ασκήσεις στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασκήσεων. Το πρόβλημα ήταν η ανταλλαγή ε, ε, εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτά τα διδάγματα που κομίσαμε. Αλλά σε τελική ανάλυση αυτό κερδίσαμε μέσω αυτών των μάχημων μονάδων. Πρώτα απ' όλα μια ισχυρή φωνή των, ε, τεσσάρων του Βίσεγκρατ και της Ουκρανίας. Συνέργεια στις δράσεις, ασφάλεια στην περιοχή, αυξημένη. Ταυτότητα στην περιοχή μας και φυσικά βελτιώνουμε τη συνοχή και ε, το κοινό πνεύμα και προωθούμε την περιφερειακή συνεργασία. Τώρα λοιπόν η Πολωνία από τον Ιούλιο πέρυσι μέχρι τον Ιούνιο φέτος έχει την ε, εναλλακτική προεδρία και από στρατιωτική άποψη συμβαίνουν τα εξή θεωρητικά. Αυτά θα θέλαμε να επιτύχουμε. Ανάπτυξη βασικών αμυντικών δυνατοτήτων για τη δική μα περιφερειακή ασφάλεια, πρακτική συμμετοχή σε πρωτοβουλίε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφάλεια τη ανατολική πλευρά και εκχώρηση δυνάμεων και ε, μέσων. Λοιπόν, α περάσουμε τώρα στην ταξιαρχία Λιθουανίας, Πολωνία, Ουκρανίας που αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα περιφερειακή συνεργασία βασίστηκε σε μια ιδέα του 2014 και τώρα μόλις πριν από δύο μέρες φτάσαμε σε πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα με την ταξιαρχία αυτή η οποία έχει έδρα στο Λούμπλιν και όπως βλέπετε στις διαφάνειες ορισμένες από τις θέσεις του διοικητή ε, και κάποιες άλλες είναι εναλλακτικέ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε διοικητή Πολωνό και μετά θα ακολουθήσει Λιθουανός ή Ουκρανός και ούτω καθεξής. Με καταμερισμό δηλαδή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων. Κλασική δομή, κάθε κράτος ε, συμμετέχει με ένα τάγμα διαφορετικού είδους ε, και φυσικά η υποστήριξη ε, γίνεται από μια χώρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση από τη δική μου τη χώρα. Συμπεράσματα, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, σχεδιάζουμε πράγματα. Φυσικά οι στρατιωτικοί πάντα κάτι σχεδιάζουν, κάτι οργανώνουν, κάτι εκτελούν. Ε, ακόμα δεν χρειάζεται να εκτελέσουμε τίποτα, να εφαρμόσουμε τίποτα. Δεν έχει παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη αλλά αν δεν σχεδιάσουμε σωστά η αποτυχία μας είναι βέβαιη. Οπότε σχεδιάζουμε διαρκώς και πρέπει να σχεδιάσουμε φυσικά μεταξύ άλλων την ε, βελτίωση της χρήσης των σημερινών εργαλείων και αυτό δεν είναι κατευθυνό όπως βλέπετε το κόστος τους αλλά φυσικά η δράση κοστίζει ε, αλλά οι δράσει μας προς το παρόν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Στρατηγέ. Ε, πολύ ας ακούσουμε τώρα τις άλλες παρουσιάσεις και μετά θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις προς το τέλος ε, του σημείου αυτού. Ε, θα δοθεί χρόνος για τυχόν ερωτήσει και απαντήσεις. Ο κύριος Ρέιτσιτς έχετε το λόγο. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σύντομη θα είναι η παρουσίασή μου και θα επικεντρωθώ στο θέμα της συνεργασίας για το V4 και, την, ε, και το τάγμα Λιθουανίας, Πολωνίας ε, και Ουκρανίας. Mm -hmm. yeah.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 στην Βαρσοβία λοιπόν είδαμε ότι σύντομα η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στις δικές της χερσαίες δυνάμεις ό,τι αφορά την προστασία της κυριαρχίας της. Σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον ασφαλείας της τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνει την Ουκρανία να αυξήσει τη συνεργασία με περιφερειακές οργανώσεις και χώρες εταίρους από, τα και, από τη Βόρεια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Γεωγραφικά ε, πιο κοντά σε αυτές τις, ε, είναι πιο κοντά αυτές τις, ε, τους οργανισμούς της Ουγγρανίας είναι το Visegrad 4, όπως λέγεται. Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Τσεχία δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας το V4, εκτιμήσαμε φυσικά την ιστορική ενότητα του οργανισμού για την υποστήριξη της Ουκρανίας από την κλιμάκωση της κατάστασης μετά τις επιθέσεις της Ρωσίας στο ανατολικό, πάρτι, στο ανατολικό μέρος της Ουκρανίας και την προσάρτηση της Κρυμαίας σε αυτή την περίοδο, όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, είδαμε ότι αυτή ήταν μία από τις ε, βασικές επιτυχίες της, ε, του V4 σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας αυτής. Το 2016 και για την προετοιμασία προς το μέλλον, πρέπει να πούμε τα εξή. Η Ουκρανία θα έπαιρνε μέρος σε αυτή τη συνεργασία με 8 αξιωματούχους καθώς επίσης και με αξιοπλισμό. Δίνοντας λοιπόν τις δυνάμεις της σημαίνει στο ομάδα μας ότι, σημαίνει ότι η χώρα αυτή δεν είναι απλώς καταναλωτής παθητικός της βοήθειας της Ευρώπης αλλά σημαντικός συνεισφέρον στην ευημερία της ομάδας και της Ευρώπης. Εδώ επίσης πρέπει να πω ότι δεν είναι νέο καθήκον αυτό για μας, νέα ευθύνη, γιατί μέχρι τότε είχαμε συμμετάσχει και στην UBG Baltic ε, του 2010 όπως βλέπετε στην ε, ε, διαφάνεια, στην e UBG Hellbrook του 2011 2012 ε, στα ανατολικά της Ουκρανίας. Επίσης και το 2014 στην ομάδα Hellbrook συμμετείχαμε και το 2016. Επίσης στην e UBG, στα πλαίσια της Προεδρίας της, του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετείχαμε στο δεύτερο εξάμεινο του 2016, του προηγούμενου τους δηλαδή. Για, στις 24 Οκτωβρίου πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Στρατιωτική της Επιτροπή συμφώνησε με τις ε, δεσμεύσεις μας για την ε, e UBG Hellbrock για το 2018 και το 2020. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ε, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες για το 2016-2017 και φάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Πολωνίας να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών των τεσσάρων κρατών μελών στην ενίσχυση της συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια στις ευρωπαϊκές χώρες. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ε, συμμετοχή σε αυτές τις, στις, ομάδες σε μεγαλύτερες επιχειρήσει επιχειρήσεις και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στο μέλλον φαίνεται ότι θα υπάρξει σκοπιμότητα να υπάρξει μόνιμη συνεργασία των ε, δυνάμεων και η συνεργασία αυτή τα επόμενα χρόνια θα, ε, θα, θα χρησιμοποιήσει συγγνώμη, τις δυνάμεις που υπάρχουν στα πλαίσια της ομαδας Β' V4, καθώς επίσης και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. From the Ukrainian side, we are looking for από την Ουκρανική πλευρά προσπαθούμε να δούμε δυνατότητες συμμετοχής της Ουκρανίας έτσι ώστε να αναζωογονωθεί η περιφερειακή συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας Βίσσεγκρατ. Καταρχάς, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα της ε, ε, ασφάλειας ε, και για την Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, δίνοντας και τις μακρόπνοες προσδοκίες της Ουκρανίας για το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια περιφερειακή δυνατότητα συνεργασίας, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τις τοπικές δυνατότητες της Ουκρανίας για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την εδαφική κυριαρχία. Αυτό θα συμβάλλει στο να αποτρέψει από τη Ρωσία να, ε, ε, χρησιμοποιήσει όλη της την ε, δύναμη και επίσης είναι σημαντικός παράγοντας να αποτρέψουμε την, την Ρωσία να επαναμοιράσει την Ευρώπη σε ζώνες επιρροής της και μη. Βεβαίω αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι θα υπάρξει συνεργασία και από την Νότια Ευρώπη και από τι υπόλοιπε χώρε στον τομέα τη ε, ασφάλεια και τη ε, άμυνα. Ο πολιτικό διάλογο επίση θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά και να θεσμοθετηθεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ε, ε στρατιωτικής ηγεσία ε, από την πλευρά της ε, Ουκρανίας για να συμμετάσχει μόνιμα στην ομαδα β V4. Τακτικές συναντήσεις με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και με τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και με τους εταίρους tv 4 έχουν γίνει πια παράδοση και πραγματικά λειτουργούν πολύ καλά. Επίσης είναι, η, σημαντική είναι η προτεραιότητα του Β4 την Ουκρανία για συνεργασία σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Επίσης ε, υπάρχει θέληση να διευρυνθεί το πλαίσιο αυτό ώστε να υπάρξει συμμετοχή και από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και άλλες χώρες. Επίσης, ε, να αναφερθώ ε, ε, στην στρατιωτική συνεργασία για να αυξηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών. Διδάγματα τώρα από τις ενόπλες δυνάμεις της ΒΙΤΕΣ και των άλλων χωρών ε, σημαίνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες κατάρτισης, ε, ε, διοικητικές δυνατότητες, κατάρτιση των στρατιωτικών, καθώς επίσης και ενίσχυση των στρατιωτικών σχολών και στα πλαίσια των χωρών 4 και στα πλαίσια των υπολείπων κρατών μελών. Επίσης, τα κέντρα αριστείας του ΝΑΤΟ αλλά και ε, κέντρα εκπαίδευσης ό,τι αφορά τις, τις ε, ε, ένοπλες δυνάμεις και την αεροπορία. Χρήση των ειδικών δυνάμεων, επίσης επιχειρήσεις ψυχολογικές, ψυχολογικού προφάιλ, η υποστήριξη των ε, ε, χερσαίων δυνάμεων είναι μερικές από τις ε, προσδοκίες μας. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία σε αυτούς τομείς έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, κοινέ επιχειρησιακές δράσεις. συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην EUBG που μπορεί να γίνει υπό την αιγίδα του, της V4 σε περίπτωση που βεβαίως αυτό ζητηθεί. στρατιωτικός εξοπλισμός, ε, προτάσεις ε, για την βελτίωση και τον εξοπλισμό των ε, όπλων είναι σημεία που επίσης θέλουμε να προωθήσουμε. Συμμετοχή της Ουκρανίας και των εταιριών της Ουκρανίας για τη δυνατότητα συντήρησης των όπλων. Στα πλαίσια του V4, της ομάδας V4, ανταλλαγή τεχνολογίας, προγραμμάτων κλπ. Πέραν αυτού, η Ουκρανία έχει εμπειρία σε συνεργασία με την Ουγγαρία και την Τουρκία εντός προγραμμάτων του ΝΑΤΟ, ε, οπότε υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Βεβαίως υπάρχει και η ε, κοινή πρωτοβουλία για τις ε, αεροπορικές δυνάμεις της Β4. Υπάρχει δυνατότητα να εξυγχρονιστούν, να εξυγχρονιστεί ο εξοπλισμός και τα όπλα της Σοβιετικής περίοδου και η επέκταση της, των δυνατοτήτων της Ουκρανία σχετικά. Υπάρχει αρκετή εμπειρία που πετέυθηκε τη διάρκεια της εφαρμογής αυτών των project, οπότε τα πράγματα προχωράνε όχι όσο γρήγορα θα θέλαμε και είναι σε προσωρινή βάση προς το παρόν τουλάχιστον. Uh, go back a bit. Okay. Now let me uh, say a few words about uh, Litpol Utlbrig. In 2007, the heads of military departments... Το 2007 οι ε, αρχηγοί της ε, Λιθουανίας, Πολωνίας και Ουκρανίας έστειλαν μια ε, επιστολή για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεών τους Έγιναν κάποιες προτάσεις. Το 2009 είχαμε τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων ε, και λήφθη μια πρωτοβουλία για την ε, στενή συνεργασία καθώς επίσης και το φόρμα που θα γινό, ε, μέσα στο οποίο θα γινόταν η συνεργασία αυτή. Ο στόχος ήταν η δημιουργία αυτής της, αυτού του τάγματος, όπως βλέπετε, Ο στόχος λοιπόν αυτής ε, ε, ε, αυτού του τάγματο ήταν να αυξηθεί η αμοιβαία συνεργασία και, η καλύτερη, και να βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας της περιοχής. Επίσης, η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών για να χρησιμοποιήσουμε την υψηλή κατάρτιση και να επιτύχουμε καλύτερη διαλειτουργικότητα. Μετά, συμμετοχή σε συγκεκριμένες δέσμες δυνατοτήτων κοινή συνεργασία και προετοιμασία του προσωπικού, κατάρτιση, ασκήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες για να υπάρξουν, να καλύτερα αποτελέσματα. Ε, κατανομή και εφαρμογή νέων προσεγγίσεων επίσης, πρότυπα ε, προγραμματισμού, ε, καλύτερη κατάρτιση των ε, στρατιωτικών της, των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. the multinational high units Επίσης διαθετησιμότητα και τιμότητα των μονάδων στα, σε όλα τα όπλα και υποστηρικτικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στα πλαίσια επίσης του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών για τον τομέα της ασφάλειας. Με βάση και την εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη Συμφωνία των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Επίσης, η συνεργασία Λιθουανίας, Πολωνίας και Ουκρανίας κατέληξε στη συμφωνία που, συμφωνήθηκε 19, που ε, υπεγράφει 19 Σεπτεμβρίου του 2014 και η τεχνική συμφωνία υπεγράφει 24 Ιουλίου του 2015. Οι εθνικές συμβολές τώρα για, αυτό το, για αυτή τη μονάδα, τη βλέπε, τους βλέπετε εδώ στην ε, διαφάνεια και βλέπετε και τις ε, τοποθεσίες σχετικά. Ε, rotation, period of time. Μετά, η ε, εναλλαγή η κυκλική ε, αναχώρα. Βλέπετε τους αναπληρωτές, τους διοικητές των μονάδων, από ποιες χώρες προέρχονται και για ποιες περιόδους χρονικές ήταν υπεύθυνη. Κατά διάρκεια του 2015 και 2016 είχαμε 18 ε, στρατιωτικούς ε, που ε, αναπτύχθηκαν στην, στη διοίκηση και ολοκλήρωσαν διάφορες επιχειρήσεις. Ξεκίνησαν οι επιχειρησιακές δυνατότητες επίσης το 2016. 25 Ιανουαρίου ε, υπήρξε η, προ... Ε, ε, διάσκεψη και μετά προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε τις δυνατότητες κατάρτισης για το 2016 Βεβαίως υπήρξε το πρόγραμμα για τις κοινέ δράσεις που ενεκρίθη. Επίσης υπήρχαν πολυεθνικές ε, στρατιωτικές ε, ασκήσεις. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2016 ξεκίνησε η εθνική επιστοποίηση και στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ε, υπεγράφει το ε, κοινό πιστοποιητικό για την απόκτηση της πλήρους ε, επιχειρησιακής δυνατότητας αυτής της μονάδας. Για το 2017 τώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεχίζονται οι δυνατότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης. Από τις 8 στις 22 Ιουλίου 2017 θα υπάρξει συμμετοχή σε πολυμερείς πολυεθνικές ε, ε, ασκήσεις ε, στην Ουκρανία και από τις 6 17 Νοεμβρίου 2017 συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις Maple Arch στην Πολωνία. Κλείνοντας, το, η, η V4 για την Ουκρανία έχει σκεφτεί την διεύρυνση της συμμετοχή της και επίσης με συμμετοχή των, ε, της Βόρειας, Κεντρικής και, Νοτιού, και Ανατολικής Ευρώπης. Ε, συμμετοχή επίσης σε κοινέ αστι... Ε, στρατιωτικές συγνώμη, επιχειρήσεις με άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να αποτελέσει μια καλή πλατφόρμα για να ενισχυθούν οι ε, αμυντικές δυνατότητες και να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. thank Εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα... Ο Γκίντιος Καρβέλης, ε, παρακαλώ. Κύριε Σταγματάρχα. Good afternoon, Madam Chair. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Γκίντιος Καρβέλης και είμαι Λιφανός. Θα είμαι σύντομος όμως στην παρέμβασή μου, διότι πολλά τα είπαν προλαλήσαντες. Θα ήθελα να σας δώσω τη λιθανική προοπτική σε ό,τι αφορά αυτό το project. Μια προοπτική που ουσιαστικά ε, απηχεί και τις απόψεις ε, που ακούσατε ε, από τους δύο προηγούμενους, γιατί τα τρία κράτη μας συνεργάζονται από την αρχή που ξεκίνησε αυτό το project, όπως και άλλοι. Η Λιθουανία σήμερα συνεισφέρει με αξιωματικούς και όπως σας είπα έχουμε έναν διοικητή και αστυνομική, στρατιωτική αστυνομία και μια μεραρχία. Από λιθανικής πλευράς εντάσσουμε τις προσπάθειές μας στην ανατολική εταιρική σχέση και θέλουμε να παράσουμε πρακτική υποστήριξη στις ουκρανικές προσπάθειες τη μεταρρύθμιση του στρατιωτικού τομέα. Η συμμετοχή της Ουκρανίας ενισχύει τη δυνατότητά της και τη σχέση της με τη Δύση και βέβαια δίνει πρόσβαση και βελτιώνει την εφαρμογή των προτύπων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αποφάσεων, διαδικασίες εκτέλεσης, βελτιώνει επίσης και τις γλωσσικές γνώσεις, στα αγγλικά. Η Ουκρανία έτσι και το στρατιωτικό της προσωπικό μπορούν να συνεργαστούν με εταίρους σε επίσης σε ένα πολυεθνικό ε, περιβάλλον. Πρακτικά θεωρούμε ότι πρέπει ε, να έχουμε ε, τα τάγματα και τις μεραρχίες σε επιχειρησιακή κατάσταση, να μπορούν στρατηγικά και τακτικά να συνεργάζονται και ενισχύεται σίγουρα και η δυνατότητά μας να δρούμε σε διεθνή περιβάλλοντα. Τώρα, πώς βλέπουμε την ανάπτυξη του προγράμματος στο μέλλον, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, όταν ε, η μεραρχία μας φτάσει να μπορεί να ε, είναι επιχειρησιακή, το 2017 θα πρέπει, πιστεύω, η ταξιαρχία, συγγνώμη, να μπορεί να προσφέρει και άλλες ε, υπηρεσίες. Πιο αργά να τα λέτε, λέει η Πρόεδρος. Επίσης όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις από την Ουκρανική πλευρά σε ό,τι αφορά το στρατηγείο και τα λοιπά θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε επίπεδο τάγματος σε ασκήσεις εκπαίδευση προσωπικού με βάση τις ουκρανικές απαιτήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα επιχειρησιακή ανάπτυξη ε, της ταξιαρχίας ε, σε διάφορες διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις. Η Λιθουανία ε, έχει επιφυλάξεις, αλλά είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να συζητήσει την ενδεχόμενη χρήση των, της ταξιαρχίας σε κάποιες αποστολές και επιχειρήσεις και σε αποστολές και πα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας την πολύ σύντομη παρέμβαση μου να πω ότι συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα απόδοση και θα συνεχίσει η Λιθουανία να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στο project. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και είμαι έτοιμος να απαντήσω ερωτήσεις όπως και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή ουσιαστικά επί Σλοβακικής Προεδρίας είχαμε προετοιμάσει το θέμα αυτό της μεσικής διάταξης. Για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Έρη Χρέχους, αν το προφέρω καλά το όνομα του συνταγματάρχου, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω κάποιες πτυχές από του σημαντικού πολύ, σημαντικού πολύ ε, Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες στις παρουσιάσεις τους, Έχουμε αυτή την συνεργασία στην Κεντρική Ευρώπη και συνεργαζόμαστε επίσης και με την Ουκρανία. Θα ήθελα να σας δώσω την εικόνα, τη σλοβακική ε, έποψη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η συμμετοχή της Σλοβακίας ε, στο UBG, δηλαδή σε αυτέ τι μάχημες ομάδες, ε, ήμασταν δραστήριοι από την αρχή. Η Σλοβακία συμμετείχε στις τρεις μάχημες μονάδες μέχρι σήμερα. Πρώτη το 2009 με τη Τσεχία ως ε, κράτος πλαίσιο. Το 2010 με Πολωνία ως σχέδιο, ως ε, χώρα πλαίσιο και συμμετοχή άλλων χωρών όπως ήταν η Γερμανία και το 2016 μαζί με την Ουκρανία και άλλες τέσσερις χώρες. Ό,τι αφορά τη συνεργασία για το 2016 το V4 και το BC, τέσσερις χώρες δηλαδή και η Ουκρανία. Θα ήθελα να πω ότι η ιδέα αυτή για τη δημιουργία κοινή μάχημη ομάδα χρονολογείται πριν από μια δεκαετία. Τελική απόφαση για τη δημιουργία αυτή τη μάχημη μονάδα το πρώτο εξάμεινο του 2016 ελήφθη το 2011. Μετά οι τέσσερι χώρες, V4 και η Ουκρανία, ξεκίνησαν συναντήσεις ε, για το σχηματισμό αυτής της ε, μάχημης μονάδας. Στη φάση της προπαρασκευής είχαμε και πολλές δραστηριότητες εκπαιδευτικές, ε, συναντηθήκαμε σε όλες τις χωρες δ V4. Η εκπαιδευτική φάση υποδιαιρεί το σε 12 τμήματα εθνικά και είχαμε και ένα εξάμεινο διεθνές. και στην Κρακοβία έγινε ε, στην Πολωνία συγκεκριμένα η τελευταία φάση της ε, εκπαίδευσης. Να σας δώσω κάποιες προοπτικές για τη μελλοντική συνεργασία V4, V4. Ήδη ξεκινήσαμε να εξετάζουμε άλλες δυνατότητες για τη μελλοντική αξιοποίηση της μάχης αυτής της ομάδας χωρίς του Βίσεγκρατ. Θέλουν να δημιουργήσουν επίσης μια κοινή μάχη με για το δεύτερο εξάμεινο του 2019. Έχει ανακοινωθεί αυτό στα επίσημα βήματα συζήτηση. Είναι φιλόδοξο αυτό το σχέδιο και ελπίζουμε να το πραγματοποιήσουμε. Πριν από αυτό όμως συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη δύο κοινά project. Το πρώτο, εκπαίδευση και στρατηγική ασκήσεων για το μέλλον και το λεγόμενο modular forces, δυνάμεις που μπορεί να διαμορφωθούν ε, σε διαφορετικά σχήματα. Θέλουμε να έχουμε ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις ως V4 για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ξεκινήσαμε να προγραμματίζουμε τον κύκλο από το 2016 στο 2020. Ένας τετραετής κύκλος λοιπόν έχει ξεκινήσει. Και έχουμε και το visibility exercise. Σε αυτά τα modular forces, που είναι το δεύτερο project, αυτό είναι σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση είναι υπέρ αυτού του προγράμματος. Θα μελετήσουμε όλες τις δυνατές εναλλακτικές για να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το project. The required state. Τέλος, ο βασικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε δυνατότητες έγκαιρης ανταπόκρισης στο πλαίσιο του V4 και πάντα των Modular Forces. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ζεσμές που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα οι δυνάμει μας θα δώσουν τη δυνατότητα κοινή δράση και ανάπτυξη ε, των δυνάμεών μα. Και για τι τρέχουσε και για τι μελλοντικέ επιχειρήσει αντιμετώπιση διαχείριση κρίσεων. Αυτά έχω, αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very... Ευχαριστούμε πολύ, αξιότιμη κύριε. Λοιπόν, προφανώς ε, πρώτος θέλει να μιλήσει ο αντιπρόεδρος της Υποεπιτρεπής Ασφάλειας, ο Γιάρομερ Στέτινα, την Τσεχική Δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, που υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ των μάχημων μονάδων της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα η συμμαχία αυτή είναι πολύ σημαντική. Ειδικότερα καθώς η Ρωσική Ομοσπονδία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την Ουκρανία. Και έχω μια πρακτική ερώτηση αξιότιμη. Ε, κύριε Συνταγματάρχη και προς τα άλλα μέρη του πάνελ μιλάτε για επιχειρήσεις που οργανώνεται από κοινού, τα κτλ. Όλα αυτά διεξάγονται και στην επικράτεια της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Uh, I, encourage uh, uh, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να συμμετέχουν στη συζήτηση και στο μεταξύ θα μπορέσουν να απαντήσουν τα μέλη του πάνελ σε αυτή την ερώτηση την οποία επιθυνέ ο συνάδελφος σε όλους σας, οπότε ένας γρήγορος γύρος απαντήσεων. Thank Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι φυσικά γίνονται κάποιες ασκήσεις, εκπαίδευση, κάποιες ε, ε, συναντήσεις, διασκέψεις, αλλά δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κανέναν και αυτό είναι το πρώτο για πολύ την προτεραιότητά μας. Όπως γνωρίζετε, η ταξιαρχία αυτή Λιθουανίας, Πολωνίας και Ουκρανίας ε, ε, υποστηρίζει και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων εφόσον το ζητήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και βασική αρχή εδώ είναι ότι αν οι γειτονέ μας ε, είναι πιο σταθεροί, τότε είμαστε και εμείς πιο ασφαλείς. Και φυσικά οι ασκήσεις αυτές γίνονται σε διάφορα εδάφη εντός των χωρών Βίσεγκρατ ε, αλλά και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία παρήχε στρατηγική μεταφορά ε, σε αυτή την περίπτωση γιατί είχα τέτοιο περιθώριο. Όπως είπαμε λοιπόν όπως είπα και οι συναδελφοί μου αναπτύσσεται και τώρα μετά από την εκτύπωση των πλήρων δυνατοτήτων προετοιμάζουμε το πρόγραμμα ασκήσεων το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την Ουκρανία σε μια λογική ε, κλίμακα. Ευχαριστώ. Κύριε Ρέιτσιτς, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εκτός μικροφώνου ο κύριος ε, ομιλητής. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα απόλυτα την ερώτησή σας. Ε, ε, δεν προέλαβα να ακούσω το διερμηνέα. Επαναλάβετε παρακαλώ. Λοιπόν, ε, επεσήμανα το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των στρατιωτικών δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας και ρώτησα κατά πόσο οι εκπαιδεύσεις που αναφέρθηκαν έλαβαν χώρα επίσης και στην, σε εδάφη της Ουκρανίας. Αυτό ρώτησα. Για να ευχαριστήσω τον κύριο ε, στρατηγό για την απάντησή του. Ευχαριστώ. Παρά την κατάσταση που έχουμε στην Ουκρανία, υπάρχει πλήρη συνεργασία με τους εταίρους μας. στις στρατιωτικές ασκήσεις και στις προετοιμασίες λοιπά Και θα διεξάγουμε ασκήσεις μαζί όταν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες και στην Ουκρανία. Έχουμε και το δικό μας εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή του Λβόβ. Και όπως εξήγησε για το 2017 έχουμε προγραμματίσει ασκήσεις και στις χώρες των εταίρων μας επίσης. Πέραν αυτού, πραγματοποιούμε διαφόρων ειδών ασκήσεις για την εκπαίδευση των εθνικών μας ε, δυνάμεων σύμφωνα με τα εθνικά μας σχέδια. και κάποιες ασκήσεις προετοιμασίας του στρατιωτικού μας προσωπικού για συμμετοχή σε αποστολές αργότερα επίσης. Ευχαριστούμε ε, συνταγματαρχή Καρβέλης, ε, θέλετε να πείτε κάτι. Είναι λίγο δύσκολο να είσαι ο τρίτος ομιλητής πάντα, ξέρετε. Ναι, λέει η Πρόεδρος, συμφωνώ και εγώ. Ε, έχω να επαναλάβω τα ίδια. Ναι, πράγματι, οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα σε όλες τις χώρες. Ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κύκλος ασκήσεων. Προηγήθηκε τώρα προετοιμασία και τώρα έχουμε στηθεί στα πόδια μας και οι ασκήσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες και κάποιες ασκήσεις, το επικυρώνω και εγώ, ε, λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστούμε κύριε Φέχος. Επικυρώνω και εγώ να, να πω δύο πράγματα. Όχι μόνο οι τέσσερις του Βίσεγκράτ και ε, στην ταξιαρχή αυτή, αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχει και συνεργασία διμερής. Σλοβακία, Ουκρανία για παράδειγμα, Πολωνία, Ουκρανία για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες διμερείς ε, συνεργασίες που προετοιμάζουμε. Να προσθέσω κάτι για τις διμερείς συνεργασίες. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με αυτή το τάγμα, ξέρετε, με τις ε, τέσσερις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Θα σας ενημερώσω. Ήθελα να σας ενημερώσω όλους ότι από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου η αποστολή της ΣΕΝΤΕ ε, ε, θα επισκεφθεί την Πολωνία στο Στσέτσιν και στη Βαρσοβία, Βαρσάβα. για να συναντηθεί με τους εκπροσώπους ε, που συμμετέχουν στην ενίσχυση της ανατολικής πτυχής του ΝΑΤΟ στις περιφερειακές προσπάθειες ε, και θα φωσιώσουμε και κάποιο χρόνο στην πολωνική, λιθουανική, ουκρανική ταξιαρχή. Αυτό θα αποτελέσει και μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε την όλο και στενότερη συνεργασία στην περιοχή μεταξύ των διαφόρων κρατών σε ποικίλε μορφές. Αυτό θα μας βοηθήσει ε, να αντιδράσουμε κάπως στις ε, ανησυχίες που εκφράζονται μετά από τις συνεχείς αυξημένες απειλές ε, που νιώθουμε από κοινού μετά από το 2008 θα έλεγα. Όπως για παράδειγμα ο πόλεμος στη Γεωργία αλλά και ειδικότερα μετά από την παρανομή προσάρτηση της Κρυμαίας ε, και την επίθεση στην Ουκρανία. Προετοιμαστήκαμε και είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα καταφέραμε να χτίσουμε τη στρατιωτική πλατφόρμα συνεργασίας με την Ουκρανία. Κύριε Στετινά, κύριε Αντιπρόεδρε, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δράτε με τις ευκαιρίες, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Είστε στρατιωτικοί αξιότιμοι κύριοι, είστε στρατιώτες και ε, πρέπει να ρυθμίσετε τα στρατιωτικά προβλήματα. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτά που κάνετε, αυτή η προετοιμασία, αυτή η συνεργασία ε, στο πλαίσιο αυτών των μάχημων μονάδων είναι μια πολιτική πράξη και θέλω να σας ευχαρώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Όπως γνωρίζετε το ε, meeting αυτό μεταδίδεται στο διαδίκτυο και μπορεί κανείς να το δει και σε αναμετάδοση στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα να σας δουν και εξωτερικοί παρατηρητές. Θα θέλατε να πείτε κάτι για να κλείσετε με πολύ σύντομη ε, μια πολύ σύντομη δήλωση. Για να μην έχουμε την ίδια σειρά, θα αλλάξουμε. Βέρι Ρέχους, ε, παρακαλώ και σταγματά, το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Καταρχάς, θέλω να πω και εγώ ότι ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέτσινα για αυτό που είπε. Ήταν πολύ ευγενικά τα λόγια του για μας τους ε, στρατιωτικούς. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία στην Κεντρική Ευρώπη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως για τη Σλοβακία. 5 εκατομμύρια. Μικρή χώρα, όπως γνωρίζετε. Χρειάζεται η συνεργασία τη χώρα μα με άλλε χώρε τη Κεντρική Ευρώπη και είναι σημαντική η συνεργασία αυτή και για έναν άλλο λόγο. Γιατί έχουμε ρίζες ε, που μας συνδέουν με την Πολωνία, με την Ουγγαρία. Το δυναμικό της συνεργασίας λοιπόν είναι πολύ μεγάλο και βασίζεται στις ρίζες μας, στην ιστορία μας. η συνεργασία στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει και για τη συνεργασία με άλλες χώρες ή μεταξύ άλλων χωρών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ασφάλειά μας και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το project για τη Λιθουανία. Η Λιθουανία από την αρχή ήταν του βασικού υποκινητέ για να ξεκινήσει αυτό το project, να γίνει επιχειρησιακό. Είναι σημαντικό για εμάς από κάθε οπτική γωνία, πολιτική και στρατιωτική, διότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα στρατιωτική συνεργασία που τελικά βελτιώνει την περιφερειακή συνεργασία, ασφάλεια και τη σταθερότητα. Όχι μόνο στην περιοχή αυτή, αλλά και, στα, ε, και πέραν των συνόρων μας. Ε, η Ουκρανία ε, είναι επίσης ένα σημαντικό σύμμαχος. Η Λιφανία θα παραμείνει ε, πιστός εταίρος αυτό το project. Ευχαριστώ. Ο συνταγματάρχης Ρέιτσιξ. Having experience Έχω εμπειρία ε, από το πώς, μπορεί πώς αντιμετωπίζει κανείς την πράξη έναν εχθρό. Και έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι καλό και για τη χώρα μας και για όλους. Η συμμετοχή σε αυτή τη ε, μάχη μονάδα, V4, Είναι κάτι που το αποφασίσαμε, όπως συμμετέχουμε και σε άλλες επιχειρήσεις και υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ αλλά και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Διότι είναι πολύ σημαντικό η χώρα μας να έχει εταίρους. Έτσι μπορούμε να προασπίσουμε τη χώρα μας από τις απειλές που δεχόμαστε. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Και ο, γενικό, ο στρατηγός ε, Φαλκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση της, ε, ε, που μας απευθύνεται στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ συζητούμε σε πολιτικό επίπεδο, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η κατανόηση. Η Πολωνία ακριβώς εκεί είναι προσανατολισμένη. Στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Και όπως είπαν, οι γείτονες μας είναι σταθεροί και εμείς είμαστε πιο ασφαλείς. Άρα θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και θα αναλάβουμε όλες τις πρωτοβουλίες για να είμαστε όπως ε, το ΝΑΤΟ. Όλοι για όλους, όλοι, ένας για όλους και όλοι για έναν. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Η Ευρώπη είναι γενός ασταθής ήπειρος και θα πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο ε, παρελθόν. Αν θέλεις την ε, ε, ειρήνη, προετοίμαζε τον πόλεμο, λέει το ρητό. Αλλά εμείς θέλουμε να πούμε και το άλλο, ότι αν θέλουμε να προετοιμάσουμε την ειρήνη, πρέπει να προετοιμάσουμε την ειρήνη. Ολοκληρώνουμε λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, και αυτό το σημείο της διάταξης και εκ μέρους όλων των μελών της υποπιτροπή Άμεσης και Ασφάλειας θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα διακεκριμένα μέλη. Το διοικητή Φαλκός και το συνταγματάρχη Ρέκη, τον ε, συνταγματάρχη Ρέχους και το συνταγματάρχη Καρβέλης. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να έρθετε και στο μέλλον να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο της συνεργασίας ε, των χωρων ΒΙΦ V4 με την Ουκρανία. Και συνεργασία Πολωνίας, ε, Λιθουανίας, Ουκρανίας, αυτή την ταξιαρχία. Και συγγνώμη που βάλα την Πολωνία πρώτα, αλλά είμαι από την Πολωνία. Να δώσω τώρα το λόγο στον Γιάρο Στετσίνα, να του δώσω την Προεδρία. Σας ευχαριστώ που ήρθα, ήσασταν εδώ αύριο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία και σας προσκαλώ θερμά.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

Good evening, ladies and gentlemen. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως με το σημείο 13, το μέλλον των μάχημων μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε περίπου μία ώρα, στους λίγο λιγότερο, και θα ήθελα να καλωσορίσω τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας τον κύριο Νίκλα Νοβάκη από το Πανεπιστήμιο του Μπερντίν, επισκέπτη ερευνητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, στο VUB των Βρυξελών, στο Φλαμανδόφωνο ε, Πανεπιστήμιο και τον ταξιάρχο Ντανιέλ Γραμμάτικο διευθυντή επιχειρήσεων, στρατιωτικό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε πιστεύω να ξεκινήσουμε αμέσως ε, τη συζήτησή μας. Έχετε τον λόγο, κύριε Ταξιάρχε. Ευχαριστώ πολύ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις ευρωπαϊκές μάχημες μονάδες για περίπου 10-15 λεπτά το πολύ. Και ουσιαστικά το θέμα, αν το θυμάμαι σωστά, ήταν το μέλλον των μάχημων ε, μονάδων. Έχω σταδιοδρομία άνω των 35 ετών στο στρατό και στο στρατό δεν προγραμματίζουμε τίποτα για το μέλλον. Αντί να σας πω λοιπόν ποιο θα είναι το μέλλον των μάχημων μονάδων, θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποια ένδειξη του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι μας προβληματίζει, τι μας απασχολεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις μάχημες μονάδες και μιλώντας για το μέλλον φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να με ξανακαλέσετε μέσα στους επόμενους μήνες ε, αν θέλετε περισσότερες διευκρινήσεις για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι το μάχημα Μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πλήρως επιχειρησιακή από το 2007. Όπως διευκρινήθηκε την αναθεωρημένη έννοια του 2015 της Ευρωπαϊκής Απόκρισης. Αυτό σας το λέω για να εξηγήσω ότι δεν είναι μια σταθερή έννοια αυτή, είναι μια εξελισσόμενη έννοια και την προσαρμόζουμε μόλις αυτό καταστεί απαραίτητο. Πρέπει όμως να πούμε ότι παρά το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα αυτής της έννοιας, οι μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καμία επιχείρηση που, της οποίας ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που ξεκίνησαν. Στη συνέχεια της ε, Ευρωπαϊκής ε, Καθολικής Στρατηγικής που πιθανότητα θα έχετε ακούσει, το σχέδιο υλοποίησης για την άμυνα και την ασφάλεια ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να επανεξετάσει την έννοια των μαχημών μονάδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προσπαθήσει να βελτιώσει ε, τι δυνατότητε ανάπτυξη των μαχημών μονάδων. Θα επανέλθω σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει επίσης να σημειώσετε ότι ανανεώνεται λοιπόν διαρκώς αυτή η έννοια, αλλά από στρατιωτική άποψη πρέπει να σας πω ότι θα χρειαστεί να βρούμε κάποιους τρόπους ε, για την εξέλιξη αυτής της έννοιας, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με τις εμπειρίες μας, τη δική μου εμπειρία ως διευθυντή επιχειρήσεων, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ε, αναπτύσσουμε τόσο συχνά στις μάχημες μονάδες ε, δεν είναι ε, η έλλειψη καταλληλότητας αλλά κυρίως για λόγους οικονομικούς και ενδεχομένως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Και για να είμαι ειλικρινής, εμείς ως στρατητικοί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα από αυτή την άψη. Οπότε η μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν πιθανότατα οι πιο, πλέον εξέχουσες ε, μονάδες ταχείας ε, παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία για το τι είναι μια μάχημη μονάδα. Είναι μια πλήρως εκπαιδευμένη, πλήρως, ε, πλήρων δυνατοτήτων μονάδα που πληρεί τα ακριβή κριτήρια όπως έχουν σχεδιαστεί. Είναι 1.500 ε, άνθρωποι ε, διαθέσιμοι ανά μονάδα που μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορα υποθετικά σενάρια που θα καλύψω αργότερα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να αναπτυχθεί εντός πέντε ημερών μετά από την ε, ειδοποίηση κινητοποίησης που είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτές οι μαχημές μονάδες ε, έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν αναφερθεί στον προσδιορισμό και που συμφωνήθηκαν από τη χώρα πλαίσιο της μάχημης μονάδας και από τις χώρε χώρες των διαφορών μάχημων μονάδων. Λόγω του μικρού μεγέθους αυτών των μονάδων είναι προφανές ότι δεν μπορούν να καλύψουν σε όλες τις περιπτώσεις ε, τις απαιτήσει ε, ε, της κάθε Οπότε, όπως και με τις άλλες επιχειρήσεις, έχουμε μια διαδικασία δημιουργίας των επιπλέον δυνατοτήτων που χρειάζονται πριν να κινητοποιηθεί η μονάδα εφόσον χρειαστεί. Το χρονοδιάγραμμα ε, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού είναι πολύ πιεσμένο όσον αφορά μια μάχημη μονάδα σε σχέση με τις κανονικές επιχειρήσεις. Αλλά βάσει της εμπειρίας μου και πάλι, δεν είναι ο χρόνος που χρειάζεται η διαδικασία σχεδιασμού το πρόβλημα, αλλά ε, η διαδικασία λήψης απόφασης και πάλι. Για παράδειγμα, ήδη γνωρίζουμε τι είναι αυτό που καθυστερεί τα πράγματα και ενδεχομένω να καθυστερεί το χρόνο που εμείς μπορούμε να κινητοποιήσουμε μια δύναμη. Ε, τι είναι, είναι φυσικά η απόφαση έναρξη της επιχείρησης αλλά και στη συνέχεια η, ο καθορισμός ενός ανατού διοικητή. Ε, I, am interacting uh, very often with the different Πολύ συχνά συνομιλώ με τις διάφορες μέχμες ε, μονάδες που έχουμε από τα διάφορα κράτη-μέλη και συνεργαζόμαστε και είναι πανέτοιμες ε, για ανάπτυξη όλες. Οπότε αυτό πρέπει να βελτιωθεί στον τρόπο ανάπτυξη των μονάδων. Δεν είναι η εργασία σε αυτές τις τρεις διαστάσεις. Ίσως γνωρίζετε επίσης, και αυτό θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, Θα ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, είχε αναλάβει μέσω του σχετικού σχεδίου ε, για την ασφάλεια και την ε, άμυνα. Τη ανατέθηκε να δώσει κάποια πρόταση για την ενίσχυση τη χρησιμότητα και τη αναπτυξιμότητα των μάχημων μονάδων, μεταξύ άλλων. Οπότε το θέμα είναι να δούμε την μορφή των μάχημων μονάδων και να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη κατά την αρχική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εργασίες, διότι όπως το καταλαβαίνω εγώ, διαβάζοντας αυτά τα λόγια και αυτά τα καθήκοντα, υπάρχει ένας κίνδυνος παρανόησης του άρθρου 10, όπως το βλέπουμε εδώ, του σχεδίου υλοποίηση. Διότι κατά βάση θα μπορούσε κανεί να καταλάβει ότι του ζητείτε να χρησιμοποιεί καλύτερα, να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιεί καλύτερα τι μαχημένε μονάδε. Ε, που σημαίνει και πάλι ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τη μάχημη μονάδα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουμε και ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζουμε την ανάπτυξή της είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε τελικά τη μάχημη μονάδα. Αλλά τελικά δεν είναι αυτός ο λόγος όπως σας είπα. Ε, this... Η αναθεώρηση αυτής της έννοιας έχει ήδη ξεκινήσει, όπως είπα στην εισαγωγή μου. Το θέμα είναι η παροχή επιμέρους μονάδων ε, βάσει δυνατοτήτων συγκεκριμένων ε, για λόγους ενίσχυσης ή προσαρμογής ε, μιας μαχημής μονάδας ανάλογα με τις περιστάσεις, την κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει. Έλεγα ότι πέρα τις προσπάθειες βελτίωσης της ευελιξίας των μαχημών μονάδων μας και ειλικρινά μπορούμε ε, διαρκώς να ε, βελτιώνουμε την ευελιξία. Υπάρχουν και άλλες οδοί, πιθανότατα. Η πολιτική βούληση για συλλογική απόφαση ανάπτυξης της μαχημής μονάδας, η χρηματοδότηση της μαχημής μονάδας, θα κάνω και μια σύντομη παρουσίαση για την πτυχή χρηματοδότησης αυτών των περιπτώσεων ανάπτυξης της μαχημής μονάδας και επίσης και το επίπεδο κινδύνου, η επικινδυνότητα. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να θέτουμε στα κρατημέλη πριν την ανάπτυξη, γιατί μια από τις αποστολές της μάχημης μονάδας είναι να αναπτύσσεται ως πρώτη ε, δύναμη. Δηλαδή η πρώτη μη τοπική δύναμη που αναπτύσσεται σε περίπτωση αναδιωμένης κρίσης, επίγουσας κρίσης ε, και φυσικά σε ένα τέτοιο πλαίσιο υπάρχει ένα επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν και να ε, αξιολογηθούν σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά τώρα αναφερόμενο στη ε, χρηματοδότηση και στην πολιτική βούληση και στο επίπεδο επικίνδυνοτητας ε, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε πολιτικά θέματα και το οικονομικό θέμα είναι πολιτικό. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη χρηματοδότηση διότι πρόκειται για ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της μάχημης μονάδας αλλά όχι μόνο, βασικά οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. παρότι παρατηρούνται κάποιες βελτιώσεις αυτή τη στιγμή ε, από αυτή την άψη. Πρέπει να ξέρετε ότι η βασική αρχή για τη χρηματοδότηση μιας ε, μάχημης μονάδας δεν διαφέρει καθόλου ε, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Ουσιαστικά, αν έπρεπε να σας πω ένα ποσό, το μόνο που θα είχα να σας πω ότι το κοινό κόστος για την ανάπτυξη μιας μάχημης μονάδας είναι περίπου το 10% τελικού κόστου της ανάπτυξης. Δηλαδή, αν ένα κράτος επιθυμεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη μιας μάχημη μονάδα, πρέπει να πληρώσει, να καταβάλει το 90% της ανάπτυξης ε, των δικών της ε, ε, στρατευμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάπω αποτρεπτικό για τα κράτη-μέλη η συμμετοχή σε μια τέτοια επιχείρηση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε παρατηρήσει ε, το τελευταίο, τον περασμένο Δεκέμβριο μία ανακοίνωση του Συμβουλίου ανέφερε ότι αυτές οι κοινέ δαπάνες θα μπορούσαν να διευρυνθούν και για την ανάπτυξη μιας μαχήμης μονάδας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του Συμβουλίου η Ειδική Επιτροπή λοιπόν για την επιχείρηση Αθηνά ε, αυτή τη στιγμή μελετά ώστε να δει πώ μπορεί να διασφαλίσει ότι η ανακοίνωση του Συμβουλίου θα μετατραπεί σε απόφαση του Συμβουλίου πρώτα απ' όλα και δεύτερον ε, προσπαθούν με την υποστήριξη των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτή την Ειδική Επιτροπή Αθηνά να συμπεριλάβουν σε αυτή την ανακοίνωση όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την επανανάπτυξη ε, και κάποια άλλα κόστη όπως ασκήσεις, ε, προπαρασκευαστικές ε, στη φάση προετοιμασίας καθώς και για την αποθήκευση όλου του εξοπλισμού που πρέπει να είναι έτοιμο πόλεμος ε, ανά πάσα στιγμή. So, uh, to, summarize... Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, εδώ βλέπετε τους διάφορους τομείς όπου μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάποια βελτίωση. Ο πρώτος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, ε, μία μάχημη μονάδα εξορισμού δεν είναι σχεδιασμένη για να αναπτυχθεί για πάνω από τέσσερις μήνες και βάσει της εμπειρία μας ε, αυτή η περίοδος των τεσσάρων μηνών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ανάγκη όσον αφορά την υλοποίηση ε, την ανάπτυξη σε ένα μη περιβάλλον σε μια χώρα που αντιμετωπίζει κάποια κρίση. Αυτό τι σημαίνει ότι μόλις αναπτύξουμε τη μάχημη μονάδα αμέσως αμέσω, μετά από την πρώτη μέρα της ανάπτυξης ήδη πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος ε, θα ηγηθεί αυτής της μαχήμης μονάδας είναι πολύ περίπλοκη δηλαδή η κατάσταση. Δηλαδή, μόλις ένα κράτος μέλος δεσμεύσει κάποια μέσα σε μια μάχη με μονάδα, ξέρουν ότι πρέπει ήδη να σκεφτούν πώς θα αντικαταστήσουν αυτούς που έχουν αναπτυχθεί επί τόπου. Ε, αυτό λοιπόν μας ε, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και μετά τίθηκε το θέμα ε, της αύξησης του αριθμού ασκήσεων, ε, αλλά αυτό δεν είναι τόσο περίπλοκο. Η επέκταση της περίοδου αναμονής επίσης είναι κάτι ενδιαφέρον γιατί μια μαχημή μονάδα αφού πιστοποιηθεί και εκπαιδευτεί ε, βρίσκεται για ένα εξάμεινο σε κατάσταση επιφυλακής και πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι όλες αυτές οι προσπάθειες εκπαίδευσης, εξοπλισμού, πιστοποίησης ε, ε, είναι κρίμα να λαμβάνουν χώρα για να Υπάρχει περίοδο επιφυλακή μόνο για 6 μήνε και η ιδέα είναι λοιπόν να επεκταθεί αυτό το διάστημα επιφυλακή σε ένα έτο ώστε να ε, αποκομίζονται όλα τα ωφέλη όλων αυτών των επενδύσεων εκπαίδευση κτλ. Και τέλο, φυσικά, μια τελευταία πτυχή για να είμαι ειλικρινής, ε, ε, πιστεύουμε ότι αυτός ο τρόπος βελτίωσης θα λειτουργήσει και να πω ότι πολύ ειλικρινά πιστεύω ότι το πιο δύσκολο θα είναι πόσο τα κράτη-μέλη τελικά επιθυμούν πραγματικά να εξετάσουν όλους αυτούς τους πιθανούς τρόπους και τομείς βελτιώσεων διότι όπως είπα βάσει της εμπειρίας μας και βάσει και της πρώτης παρουσίασης που κάναμε εμείς ε, ως επιτελείο ε, στην Στρατιωτική Επιτροπή μια, πριν μια εβδομάδα περίπου την ίδια παρουσίαση μάθαμε από τα κράτη-μέλη, ακούσαμε από τα κράτη-μέλη τόσες ε, πολλές ε, ε, διαφορετικού είδους συμβουλές και θέσεις που μερικά κράτη-μέλη είναι έτοιμα να, να αλλάξουν τελείως την όλη έννοια και άλλα δεν θέλουν να, ούτε επιθυμούν να κάνουν απολύτως τίποτα παρά να παραμείνουμε σε κατάσταση επιφυλακής όσον αφορά αυτή τη μάχημη μονάδα. Πρέπει να ξέρετε ότι η ευελιξία ε, κάτι που σημαίνει ευελιξία, δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστου περιορισμού στο σχεδιασμό. Απλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν. Αν ε, θέσουμε πολλού περιορισμού, ε, θα χάσουμε την υποστήριξη των κρατών μελών ή ορισμένων κρατών μελών. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανεί για να κλείσουμε. Μάλλον είναι προ... καλύτερο σε αυτό ο σχηματισμό από από άλλους. Είναι προτιμότερο να έχουμε ένα τελή σχηματισμό από το να έχουμε έναν τέλειο σχηματισμό χωρίς καμία συμμετοχή των κρατών. Είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ε, ερώτηση θέλετε. Ευχαριστούμε κύριε Στρατηγέ. Να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση μόλις ακούσουμε και τον κύριο Νοβάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσω για το μέλλον των ε, μάχημων μονάδων. Και, μενα μου, και εγώ περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι όντω ε, πολύ καλή χρονική στιγμή να συζητά κανεί το μέλλον των ε, μονάδων μάχη, μια που το 2017 αποτελεί και το έτο τη 10 η επαιτίου της ε, πλήρου επιχειρησιακή δυνατότητα των μονάδων μάχης. Ξεκίνησε δηλαδή το 2007 και η ευρωπαϊκή φιλοδοξία ήταν να υπάρχουν δύο μονάδες μάχης σε stand-by μόνιμα. Η επέτειος όμως αυτή βεβαίως δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα σε όλη την Ευρώπη. Και ο λόγο είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ετών που βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση, οι μονάδε μάχη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. E uh, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να θέλει να ε, αναπτύσσει ad hoc επιχειρήσεις οι οποίες ε, δημιουργούνται και συστήνονται αναπερίπτωση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβει. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα τελευταία χρόνια είδαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για αυτές τις μονάδες μάχης στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό φαίνεται και από τα από το ρόστερ που δεν είχε πληρότητα τα τελευταία χρόνια για τις ε, μόναδες μάχης. Επίσης ε, υπήρξαν ε, κάποιες σκέψεις που έλεγαν ότι ίσως έπρεπε να, να, ξανασκεφτούμε τι σημαίνει μόναδες μάχης και πώς μπορούμε όντως να τις κάνουμε πιο επιχειρησιακές. Υπήρξε η στρατηγική του 2016 καθώς επίσης και το εφαρμοστικό σχέδιο, κάτι που επανέλαβε τις ανησυχίες αυτές. Αλλά το βασικό ερώτημα που θα έπρεπε ίσως να θέσει κανείς ε, για την ανθεώρηση των ε, ε, μονάδων μάχης είναι το κατά πόσο αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα βελτίωναν την δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των μονάδων μάχης. Κατά την άποψή μου, οι προτάσεις που υπάρχουν τώρα επιτάπητος σε ό,τι αφορά το εφαρμοστικό σχέδιο για την άμυνα και την ασφάλεια, δεν θα αύξαναν σημαντικά την δυνατότητα ανάπτυξη των μονάδων μάχη, γιατί είναι τεχνικέ οι προτάσει και το βασικό πρόβλημα των μονάδων μάχη είναι πολιτική φύσεω κυρίω. Οπότε, τι προτείνετε. Η συνολική στρατηγική λέει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για άμεση απάντηση, αντιμετωπίζοντας και τα διαδικαστικά και πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που αποτρέπουν την ανάπτυξη των μονάδων μάχης και, να, και μειώνουν την δυνατότητα ε, παρέμβασης ε, των ε, επιχειρήσεων ΚΕΠΑ. Αυτό ήδη ξεκίνησε και αναφέρεται συγγνώμη και στα συμπεράσματα του 2013 του Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ότι οι μονάδε μάχη θα πρέπει να είναι πιο λειτουργικέ. Υπάρχουν λοιπόν και αρκετοί, αρκετές προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, να αυξηθεί το αξιόμαχο των μονάδων μάχης. Ε, ας πούμε, η, ε, προσέγγιση που είχαμε από την ε, η παλιά προσέγγιση που είχαμε, ε, ενίσχυση επίσης των ε, δυνατοτήτων τους και καλύτερη χρηματοδότηση. Για να δούμε πιο λεπτομερώς αυτές τις δυνατότητες. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει μια λύση για την άτεκτη δομή των μονάδων μάχης. Όταν ξεκίνησε το σκεπτικό αυτό, βασίστηκε στην επιχείρηση Άρτεμις που έγινε στην, ε, στο Κονγκό, στη Δημοκρατία του Κονγκό το 2003 για να βοηθήσουν το, τον ΟΗΕ να διατηρήσει τη σταθερότητα στην περιφέρεια του Ήτουρη. Περίπου 1500 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν για την επιχείρηση αυτή. Και όταν λοιπόν ε, υπήρξε όλη, το όλο σκεπτικό για τις μονάδες μάχης, ε, χρησιμοποιήθηκε αυτό, αυτή η άγουσα και για τις μελλοντικέ επιχειρήσεις. Αλλά είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να έχει πιο ευρύ πεδίο επιχειρήσεων, που δεν ε, σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα ακολουθούν πάντα το μοντέλο Artemis. Οπότε η ε, πολυτροπικότητα, ας πούμε, θα πρέπει να σημαίνει ότι προστίθενται δυνατότητες εξοπλισμός, στρατιωτική, στις μονάδες μάχης που δεν ήταν αρχικά έτσι φτιαγμένες. Οπότε οι μονάδες μάχης ουσιαστικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο θα βασίζονται επιπλέον μοντέλα ανάλογα με την ανάγκη της κάθε επιχείρησης κάθε φορά. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν ε, εκπονήθηκε μόλις το 2014 για να αναθεωρήσει την άμεση αντίδραση και να ενισχύσει την ε, ΚΕΠΑ. Το θέμα είναι ότι αν η δομή των ε, μονάδων μάχης ήταν πιο ευέλικτη, τότε θα μπορούσαν να, χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιηθούν σε, μεγαλύ, σε περισσότερες κρίσεις, οπότε θα μπορούσε να βελτιωθεί το αξιόμαχό τους. Βεβαίω δεν είναι εγγύηση ότι αυτού του είδου η άγουσα θα μπορέσει να λειτουργήσει, ακόμη και αν ε, όντω ε, χρησιμοποιούνταν οι μονάδε μάχη, αλλά επίση δεν είναι και κατά ανάγκη ε, θέσπατο ότι θα χρησιμοποιηθούν οι μονάδε μάχη αν υπάρξει κρίση. Επίση, ίσω οι μονάδε μάχη να μην έχουν τίποτα, κάποιο χαρακτηριστικό που να τις διαχωρίζει από τις ε, συνήθεις επιχειρήσεις ε, άμυνας και ασφάλειας. Μετά, το, ο κοινός, ε, το κοινό αποθεματικό, ας πούμε, των πόρων. Εδώ βλέπουμε έλλειψη σε επίπεδο κρατών μελών δυνατοτήτων, κυρίως στο επίπεδο των μικρών κρατών μελών. Αυτό καθεστά πολύ επαχθές για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτές τις, ομάδες, να ε, μπορέσουν να, έχουν, ε, την, ε, να, αναλάβουν το δικό τους κομμάτι. Και έτσι η ευθύνη επαφίεται στη χώρα με, πάνω σε, στην βάση της οποίας δημιουργείται η μονάδα μάχης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ένας ε, ε, κορβανάς από τον οποίο θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τους πόρους για να δημιουργήσει τις μονάδες μάχης. Και αν υπάρχει όντω αυτό το αποθεματικό, τότε η ανάπτυξη των μονάδων μάχης θα είναι πιο, πιο αυξημένη, γιατί έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθούν οι πόροι και να δημιουργηθούν οι μονάδες μάχης. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι αν δημιουργηθεί τέτοιο αποθεματικό, τότε οι δυνατότητες που θα πρέπει να έχει θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμες. Και αυτό μπορεί κάποιες στιγμές να μην είναι δυνατόν, αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη. Και για να αγγιηθεί κανείς την διαθεσιμότητά τους μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νομικά μέσα. Επίσης, αυτό το κοινό αποθεματικό των δυνατοτήτων δεν σημαίνει ότι δημιουργούνται κατά ανάγκη δυνατότητες, απλώς καλύπτει κάποιες ελλείψει των στρατηγικών μονάδων από τις οποίες υποφέρουν τα κράτη-μέλη. Μετά, κοινή χρηματοδότηση. Η κοινή χρηματοδότηση δίνει μια λύση σε αυτό το υποτιθέμενο πρόβλημα της κατανομή των βαρών για τι μοναδέ μάχης. Όπω είπε και ο ταξίαρχος, η χρηματοδότηση των μονάδων μάχης γίνεται με βάση ε, του κόστους που δημιουργείται. Ας πούμε, ε, ό,τι, χρηματο, χρηματοδοτεί το κάθε κράτος μέλος ε, το δίνει και για τις μεικτές μονάδες μάχης. Σε, ό,τι χρηματοδοτεί δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίω είναι άδικο οι χώρε που δεσμεύουν τι δυνατότητέ του για τι μονάδε μάχη και αναλαμβάνουν όλο τον κίνδυνο ουσιαστικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι μονάδε μάχη, να πρέπει να είναι αυτέ που ουσιαστικά θα αναλάβουν και την πλειοψηφία του, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστου σε περίπτωση που όντω χρησιμοποιηθούν οι μονάδε αυτέ μάχη. Οπότε αυτή η πρόταση στην πράξη σημαίνει ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή τη κοινή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού Αθηνά. Οπότε, αν υπάρξει αύξηση του κοινού της κοινή χρηματοδότηση, σημαίνει περισσότερου πόρου ε, προ χρήση των ε, μονάδων μάχης. Βεβαίω δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ κρατών μελών για την αναγκαιότητα ή την επιθυμία της ε, διεύρυνσης της χρηματοδότηση, όπως είδαμε από την αναθεώρηση του 2014-2015 του Μηχανισμού Αθηνά. Οπότε, ενώ αυτέ οι προτάσει ε, είναι επιτάπητο και θα μπορούσαν ίσως να, ε, να δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για την ανάπτυξη των μονάδων μάχη, ουσιαστικά θα μειώσουν και την ε, δυνατότητα ανάπτυξή του, κυρίω γιατί ε, οι λύσει αυτέ είναι τεχνικέ, ενώ αυτό που χρειάζεται στι μονάδε μάχη είναι πολιτική απόφαση. Ο λόγο για τον οποίο οι μονάδε αυτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τότε που άρχισαν να είναι λειτουργικέ δεν ήταν επειδή δεν υπήρχε πολυτροπικότητα ή αυτός ο κοινός, αυτό το κοινό αποθηματικό για τους πόρους ή δεν υπήρχε κοινή χρηματοδότηση αλλά κυρίω γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική βούληση είναι πάντα περίπλοκο, περίπλοκος όρος να οριστεί στην πράξη. Αλλά ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι μια πρόθεση, μια επιθυμία, δέσμευση να εφαρμόσει κανείς τις πολιτικές του ακόμη και αν δεν είναι άμεσα πολύ δημοφιλής ή επιτυχής. Από το 2005, όταν οι πρώτε μονάδε μάχη ε, κατέστησαν λειτουργικέ, τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν ακριβώ λόγω τη έλλειψη πολιτική βούληση. Για παράδειγμα, το 2006 τα Ηνωμένα Εθνή ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να, να στείλει μία μονάδα μάχη στο Κονγκό για να βοηθήσει την διατήρηση τη σταθερότητα και τη ειρήνη στη χώρα κατά τη διάρκεια των γενικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, η μονάδα που απεστάλλει ήταν γαλλογερμανική. η Γερμανία ήταν ιδιαίτερως διστακτική να στείλει τη μονάδα μάχης στην οποία συμμετείχε και κατά το μεγαλύτερο μέρος για να χρησιμοποιηθεί στις εκλογές του Κονγκό. Οπότε αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει μια, μια ομάδα μια συνήθη ομάδα αποστολή στα πλαίσια της ΚΕΠΑ στο Κονγκό. Μετά, η ε, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία η οποία ε, αντιμετώπισε διάφορε, ε, διάφορες φιλετικές διαμάχες. Εκεί είχε αποφασιστεί πάλι να ε, σταλεί άτυπα έστω μία μονάδα μάχης. Η μονάδα αυτή που βρισκόταν σε stand-by το δεύτερο εξάμεινο του 2013 ήταν αυτή που επικεφαλής της οποίας ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και για προφανείς εσωτερικούς πολιτικούς λόγους το Ηνωμένο Βασίλειο δίστασε να στείλει τη μονάδα αυτή να χρησιμοποιηθεί στην κεντρική αφρικανική δημοκρατία, οπότε δεν ε, χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Το πρώτο εξάμεινο του 2014 η μονάδα που ήταν ε, σε stand-by ήταν ε, υπό την αιγίδα της Ελλάδας. Αλλά και πάλι η Ελλάδα δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί η μονάδα αυτή, γιατί φοβήθηκε ότι μπορεί να μην θεωρηθεί δημοφιλής απόφαση απέναντι στο λαό ο οποίος ήδη είχε ξεκινήσει να κάνει περικοπές λόγω της ευρωπαϊκής κρίσης. Οπότε η πολιτική βούληση είναι σημείο κλειδί. Στο μέλλον, αυτή η πολιτική βούληση για τη χρήση των μονάδων μάχης ε, μπορεί να αυξηθεί ε, και οι λόγοι είναι οι εξής. Καταρχάς, η κρίση στην ε, ε, Ουκρανία, με την παρέμβαση της ε, Ρωσίας. Πολλοί έχουν αρχίσει να ε, επικεντρώνονται πάλι στην κλασική άμυνα των εδαφών τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενδιαφερθούν πάρα πολύ να υπεραμεινθούν ξένων χωρών ή άλλων εδαφών όπου θα χρειαστεί να αναπτυχθούν οι μονάδες μάχης. Μετά, η, τα μόνιμα αντιευρωπαϊκά αισθήματα σε όλη την υπηρεσία της Ένωση, που σημαίνει ότι πολλά κρατημέλη δεν θα σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν ε, την, ε, ή να στείλουν μονάδες μάχης σε απομακρυσμένες χώρες εάν ε, πρόκειται να θυμώσει αυτό το εκλογικό του σώμα. Τι μπορεί να γίνει τώρα. Περιορισμένες είναι οι δυνατότητε μα γιατί οι τεχνικέ αναθεωρήσει που γίνονται ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αυξήσουν το αξιόμαχο των ε, μονάδων μάχης γιατί δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την πολιτική βούληση που είναι αυτό που λείπει. Ε, σε έναν ιδιαίτερο κόσμο αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν τα κράτη-μέλη να, δημιουργήσουν, να έχουν μια κοινή κατανόηση των προτεραιοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα, έτσι ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη των μονάδων μάχης. αυτά, αυτό δεν θα γίνει γιατί οι χώρες όπως η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία πάντα θα έχουν συμφέροντα και προτεραιότητες άμυνας και security διαφορετικά από τις χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως θα μπορούσαμε να μελετήσουμε πέραν των όσων έχουν ήδη προταθεί. Το πιο προφανές και αυτό που είπε και ο ταξίαρχος προηγουμένως είναι η δήλωση αυτή για την, ε, ε, κοινή, ε, για την κοινή χρηματοδότηση που θα πρέπει να μπει στην, στο μηχανισμό Αθήνα, έτσι ώστε να προωθηθεί το θέμα τουλάχιστον της μεικτής χρηματοδότησης. Αυτό προς το παρόν μελετάτε. Αυτή η αναθεώρηση γίνεται κάθε δύο χρόνια του μηχανισμού, αλλά μπορεί κάποιε φορέ να καθυστερήσει. Έχει, ε, το 2015 α πούμε υπήρξε μια ατυχή περίσταση όπου η δήλωση δεν εφαρμόστηκε και η Nordic ε, μονάδα μάχης ε, των σκανδιναβικών χωρών που ήταν σε stand-by δεν ήταν ε, σίγουρη σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να παρέμβει αν θα, ήταν, αν θα είχε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ένα δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι η αντίθετη, αντίστροφη τροπικότητα. Αν δεν χρησιμοποιηθούν αυτές οι μονάδες αλλά είναι σε stand-by θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει κάποιες πτυχές, κάποια modules από αυτές τις μονάδες, κάποιες δυνατότητες δηλαδή που έχουν, σε, σε, σε, σε πρότυπες ε, αποστολές σε ΚΕΠΑ, για να τις ενισχύσει. Και επίσης κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να έχουμε υπόψη είναι ε, αυτό το curtain call που ονομάζω εγώ, δηλαδή οι μονάδες μάχης να, για κάποιο χρόνο να, να βγουν από το καθεστώς πλήρους ε, μάχημης κατάστασης. Υπάρχει προηγούμενο για να γίνει αυτό στο ΝΑΤΟ, όπου το ΝΑΤΟ το 2007 έβγαλε τις ε, μονάδες ε, ανταπόκρισης από, την, από το καθεστώς πλήρους ε, ε αξιομάχου μέχρι να αναθεωρηθούν οι σχετικές ρήτρε. Για να κλείσω λοιπόν, το μέλλον των μονάδων μάχης δεν φαίνεται να είναι πολύ βίωνο. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την, για την άμυνα και την ασφάλεια είναι κυρίως τεχνικές και άρα δεν θα αυξήσουν το αξιόμαχο και την δυνατότητα ανάπτυξης των μονάδων μάχης σημαντικά. Γιατί ε, αυτό που λείπει για να γίνει αυτό είναι η πολιτική βούληση. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι μονάδες μάχης είναι, μια, είναι ένα εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρξει μια κοινή κατανόηση μεταξύ των κρατών μελών του τι σημαίνουν οι προτεραιότητες ασφάλειας και άμυνας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση των μονάδων αυτών. Και επίσης ε, να σας αναφέρω κάτι από το Διεθνές ε, ε, Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών. Παραθέτω η αργή πρόοδο στον τομέα της ε, των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων ε, δεν θα είχε κανένα λόγο ύπαρξη αν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Ευρωπαίους. Αυτό νομίζω ότι ουσιαστικά έχει το... Ε, περιλαμβάνει όλο το ζουμί της υπόθεσης, κάτι που ίσχυε δυστυχώς και για τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νοβάκη. να αρχίσει η συζήτηση. Κυρία τη αντιπρόεδρε, που θέλει το λόγο. Ναι, βεβαίω, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλέρο και εγώ, αλλά μάλλον η κυρία Βαλέρο πρέπει να πάρει το χρυσό μετάλλιο για τη συνεχή παραμονή εδώ και πραγματικά είναι περίοδο ότι συζητούμε εδώ για το μέλλον των μάχημων μονάδων, ε, για νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης ε, και ούτω καθεξής, αλλά δεν φαίνεται ενδιαφέρεται κανείς για όλα αυτά. Μια παρατήρηση έχω να κάνω. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη συζήτηση για τον καιρό του post-fact. Σε ό,τι αφορά δε, την, το πεδίο, ε, την εμβέλεια ε, δράσης αυτών των μάχημων μονάδων, μπορεί και να και 5.000 χιλιόμετρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι μέσα σε 5-10 μέρες ε, να είναι επιχειρησιακές οι μονάδες. Ε, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις στην ε, Γερμανία σε ό,τι αφορά την, το αξιόμαχο, την ετοιμότητα επέμβασης αυτών των μονάδων. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα. Μέχρι και να οργανωθεί μια έγκριση από τα κοινοβούλια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ε, κράτη-μέλη και κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη πρέπει να δοθεί η έγκριση από το Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε λοιπόν τη διαδικασία αυτή γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη με ναι, την επιφύλαξη των κοινοβουλίων. Πώς μπορείτε να το οργανώσετε λοιπόν. Και στο τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Έγιναν συζητήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ. Βάλτε τα ακουστικά σας καλύτερα θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είμαστε οι φορείς λήψη αποφάσεων. Πριν έρθω εδώ βέβαια ήμουν στο Συνδικό Κοινοβούλιο που και εκεί ήμασταν υπεύθυνοι για τα χρήματα των φορολογουμένων. Και πώς χρησιμοποιούνται σε ό,τι αφορά αυτές τις μονάδες. Ξέρουμε ότι έρχονται με μια τιμή, κάτι κοστίζουν. Και παρότι κάτι κοστίζουν δεν χρησιμοποιούνται. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Και αυτό είναι το ελάττο πρόβλημα. Εγώ και άλλοι νομοθέτες που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τα δημοσιονομικά ζητήματα. Και είμαι και πράσινη. Άρα με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει οι νευνευτικές διαδικασίες, ναι, και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δεν συνεργαζόμαστε και πολύ με τον ΟΗΕ. Αλλά μπαίνουν πάρα πολλά χρήματα στον Κορβανά για αυτά ε, τα battle groups. Ε, πώς θα το εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας αυτό ότι χρηματοδοτούμε κάτι που δεν χρησιμοποιείται. Και έρχομαι σε αυτό που είπατε και εσείς κύριε Νοβάκη για την πολιτική βούληση που λείπει. Αν δεν έχουμε πολιτική βούληση πίσω από τα battle groups δεν θα χρησιμοποιηθούν. Και οι πολίτες δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πληρώνουμε κάτι που δεν το χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάτι παραπάνω από εσάς. Τι χρειάζεται να αλλάξει μπορούμε να έχουμε με ένα άλλο μοντέλο ενδεχομένως. Αν έχουμε τα battle groups και θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε για ειρηνευτικές αποστολές, ίσως ναι, αυτό είναι καλό. Αν τα έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως πολιτική βούληση και αν υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιούνται παραλαμβάνω για ειρηνευτικές αποστολές. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Όχι, δεν ολοκληρώνεται η συζήτηση. Να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ κάποιε ερωτήσει. Αλλά μην βγάλετε τα ακουστικά. Να μιλήσω κι εγώ στη γλώσσα μου, τα τσέχικα. Τρία σύντομα ερωτήματα. Ξέχασα ότι πρέπει να μιλήσω τσέχικα. Τώρα μιλάω τσέχικα. Σε ό,τι το ΝΑΤΟ είναι το πρώτο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό συζητάει τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και τακτικών μάχημων ομάδων. Έχουν κάποια σχέση με το ΝΑΤΟ, επαφή, το ΝΑΤΟ τι στάση έχει απέναντι σε αυτά. Και τι όπλα χρησιμοποιούν. Στο Κόγκο, για παράδειγμα, τι κατηγορία εξοπλισμού χρησιμοποιούσαν. Και τρίτη ερώτηση, η Ουκρανία. Την τελευταία φορά, όταν ο Ποροσέγκο ο πρόεδρος είχε έρθει εδώ στο κοινοβούλιο, μας παρακάλεσε με τεπιμονής. Μήπως θα μπορούσαν κάποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις να φροντίσουν για να κλείσει η μεθόριος Ουκρανίας ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γιατί αν τα στεγανά τα σύνορα θα έλυγε ο πόλεμος γρήγορα. Αυτοί, αυτές οι μάχημες μονάδες είτε τώρα είτε στο μέλλον θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη τις ουκρανικές μονάδες. Είναι βασικό θέμα στον τόμπας, στην Ουκρανία. Το ίδιο αίτημα θα ακούσετε. Βοηθήστε μας να στεγανοποιήσουμε τα σύνορα. Αυτά είναι όλα τα ερωτήματα. Να απαντήσετε παρακαλώ. Δεν ξέρω, στρατηγέ μου, να ξεκινήσετε. Ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να μιλήσω γαλλικά, ωραία. Και να ξεκινήσω από το πιο δύσκολο ερώτημα, το τελευταίο θα μπορούσα να κάνω έτσι ένα, μια κροβασία και να σας πω ότι είναι πολιτικό θέμα και εγώ δεν μπορώ ως ε, στρατιωτικός να επέμβω και να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αλλά δεν θα παρακάμψω τη δυσκολία και θα σας δώσω κάποια τεχνική απάντηση. Το πώς θα γίνουν στεγανά τα σύνορα. Αυτό δεν εντάσσεται σε καμία περίπτωση στις δυνατότητες στρατιωτικές ε, μιας μάχημης μονάδας. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση ενός στρατιωτικού. Εγώ θα πάω και πιο πέρα όμως και θα πω ότι αν θέλουμε να δώσουμε μια πολιτική απάντηση και θα το διακινδυνεύσω εδώ, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμμετέχει ή να παρεμβαίνει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, γιατί από τη στιγμή που θέλει κανείς να βοηθήσει την Ουκρανία, γιατί για αυτήν μιλήσατε, τότε τοποθετείται και παίρνει μέρος. Παίρνει τοποθετείται υπέρ ή κατά μιας πλευράς. Προσωπική άποψη. Για το Κονγκό, στη επιχείρηση Άρτεμις, για τον εξοπλισμό που είπατε. Δύσκολο να απαντήσω. Όλες οι μάχημες μονάδες όμως έχουν λίγο πολύ αντίστοιχο, παρόμοιο εξοπλισμό. βασικό, το βασικό εξοπλισμό ουσιαστικά. ενός είδους ταξιαρχίας. Δηλαδή δεν έχουν πολύ βαρύ εξοπλισμό και είτε ε, αποκαθιστούν την ειρήνη είτε είναι η πρώτη ας πούμε διείσδυση σε ένα δύσκολο περιβάλλον αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν. Δεν ε, υπερβαίνουν τι δυνατότητές τους. Δεν έχουν βάλει εξοπλισμό. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, θα μπορούσα να προσθέσω ότι τα battle group που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικών κατηγοριών. Κάποια έχουν πολύ ελαφρύ εξοπλισμό και κάποια άλλα έχουν λίγο πιο μεγάλες στρατιωτικές δυνατότητες όπως αυτό που έχει ως έθνος πλαίσιο την Πολωνία. Από τη θωρακισμένων, ε, από τα ξερχεία τεθωρακισμένων προβλε... προέρχεται. Και μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε 5-10 μέρες αυτά τα battle groups. Ένα άλλο είναι το Nordic Battle Group που μου έρχεται στο μυαλό. Σουηδέ, Σουηδή είναι το Framework Nation και ίσως είναι και το πιο συμπαγές, σταθερό. Έχει χερσαίο εξοπλισμό, αλλά και ελικόπτερα και γενικά αεροπορικό εξοπλισμό. Υπάρχει λοιπόν ένα βρυφάσμα σχετικά, αλλά για να απαντήσω για το Άρτεμι συγκεκριμένα, ήταν ελαφρύς ο εξοπλισμός του συγκεκριμένου τάγματος. Σε ό,τι αφορά τις 5-10 ημέρες για την ανάπτυξη που είπατε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα γιατί πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια η απόφαση. Είναι εξαιρετικό το ερώτημα. Γιατί πράγματι υπάρχει προθεσμία 5-10 ημέρες, 10 ημέρες για την ανάπτυξη του τάγματος. Άπαξ και απόφαση σε πολιτικό επίπεδο. Άρα η πολιτική διαδικασία προηγείται της ανάπτυξης της μάχης μονάδας. Και μόνο αφού ληφθεί η απόφαση από το Συμβούλιο για την έναρξη, τότε ξεκινάει η αντιστροφή μέτρηση. Άρα δεν περιλαμβάνεται στις 5-10 μέρες αυτές που σας είπα ε, το πολιτικό σκέλος. Thank you, ε, Mr. Novaki, floor is yours. Κύριε Νοβάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα των μαχημών μονάδων, είναι πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Για πολλά κράτη-μέλη που πρέπει να εγκρίνουν την ανάπτυξη των μάχημων μονάδων από τα κοινοβουλιά τους πριν εγκριθεί η ανάπτυξη. Συμφωνώ με τον ε, στρατηγό εδώ. Ε, οι επιλογές μας σε αυτό το τομέα είναι περιορισμένες. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να γίνει για να διευκολυνθεί η διαδικασία ε, στα αρχικά στάδια θα ήταν να σχεδιαστούν, να εκπονηθούν τα, οι νομοθεσίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έγκριση εκ των προτέρων ώστε να υπάρχουν έτοιμα τα έγγραφα αν έρθει η ώρα ανάπτυξης. Πέραν αυτού είναι δύσκολο να πει κανείς ε, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Δεύτερον, ε, το ζήτημα του κόστους σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ έχουμε το επίκεντρο του προβλήματος όσον αφορά τις μάχημες μονάδες και η ερώτηση είναι ε, κέρια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παρότι παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες όπως πιο πρόσφατα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ήταν ευνοϊκό το περιβάλλον για τέτοιες επιχειρήσεις Πολλοί κόσμοι λοιπόν να ρωτιέται εύλογα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτέ οι μάχημε μονάδε και για ποιο λόγο πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του. Δεν έχω κάποια καθαρή απάντηση γι' αυτό δυστυχώ. Πιστεύω επειδή ρωτήσατε κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, άλλες, για άλλους σκοπούς όπως ειρηνευτικές ε, δράσεις. Γιατί όχι. Ε, η δύναμη απόκριση του ΝΑΤΟ που είναι ένα παρόμοιο εργαλείο, λίγο μεγαλύτερο βέβαια, ε, έχει χρησιμοποιηθεί και στις Ηνωμένε Πολιτείε μετά από τον τυφώνα Κατρίνα και τις καταστροφές που προκάλεσε για ανακούφιση καταστροφών. Ε, οπότε θα μπορούσαν οι μάχημες μονάδες να χρησιμοποιηθούν και κάτι παρεμφερές παρότι αυτό θα απαιτούσε κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία για να καταστεί δυνατό. Τρίτον, κατά πόσο οι μαχημε μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία. Ο στρατηγός ήδη έδωσε μια άριστη απάντηση. Να σας πω εγώ ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα για τα κράτη-μέλη που δύσκολα μπορώ να φανταστώ μια κατάσταση όπου θα ενέκρινα να, να στείλει μια μαχημή μονάδα στην περιοχή του Νταμπάς για παράδειγμα όταν ήδη δεν εγκρίνουν την ανάπτυξή του σε μια χώρα χαμηλότερη ένταση όπω την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω σε κάποιε άλλε ερωτήσει που απομένουν. Η πρώτη αφορά την πιθανή σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μαχημών μοναδών του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Από όσο γνωρίζω εγώ δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση μεταξύ του οργανισμού τέτοια απόκριση. Ε, πέραν του ότι μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία σχεδιασμού, τον ίδιο τρόπο ασκήσεων και εκπαίδευση των διαφορών μονάδων μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν μη τι άλλο δεν συνεπάγονται όλα αυτά πρόσθετο φόρτο εργασία για τα κράτη-μέλη είναι έτοιμη δηλαδή η μαχημή μονάδα για επιχειρήσει του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι τώρα στα 22 κράτη-μέλη που ανήκουν και στους δύο οργανισμούς. Επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι λόγω του ενιαίου συνόλου πόρων και δυνάμεων τα 22 κράτη-μέλη που ανήκουν και στους δύο οργανισμούς ε, αυτό που ισχύει λοιπόν ότι όταν εκπαιδεύουμε μια μονάδα για, ως ευρωπαϊκή μάχημη μονάδα ή ως ε, ε, ομάδα ταχείας απόκρισης την εκπαιδεύουμε με τον ίδιο τρόπο εξορισμού για την πλευρά του ΝΑΤΟ. Πέραν αυτού όμως ε, δεν υπάρχει από κοινού, από ανάληψη ε, του φόρτου εργασία ε, ή οποιοδήποτε άλλο φόρτο από του δύο οργανισμού. Γίνονται συζητήσει τώρα με τα Ηνωμένα Έθνη ώστε να αξιοποιηθεί ενδεχομένω σε ειρηνευτικέ διαδικασίε του ΟΗΕ η μαχημή μονάδα. Ρωτήθηκε, ναι, πράγματι γίνονται τέτοιε συζητήσει αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε λάβει κάποιε ενδιαφέρουσε ιδέε όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη μάχημη ομάδα εφόσον εργάζεται εντό πλαισίου εντολή των ΟΗΕ. Το πρόβλημα είναι η οργάνωση επιτόπου. Διότι το, το ζήτημα τη διοίκηση τέτοιων μάχημων μονάδων σε τέτοια πλαίσια. Τα πράγματα κινούνται, αυτό πρέπει να πω. Αργά με ένα, αλλά κινούνται. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι κι εσείς. Ε, ε, ειδικότερα για το ενιαίο σύνολο ε, εξοπλισμού και πόρων. Ναι, ευχαριστώ. Για να απαντήσω στη Σουηδική, στο Σουηδικό σχόλιο, εγώ επισκεφτήκα τη Σουηδική Μάχημη Μονάδα πριν από δύο-τρία χρόνια όταν βρισκόταν σε επιφυλακή και από πολιτική άποψη ε, η Σουηδία είναι πιθανότητα ένα από τα κράτη-μέλη που έχει την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσει τη μαχημή μονάδα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, όταν μιλάμε για σπατάλη χρημάτων ε, σε περίπτωση μη χρήση τη ε, μαχημή μονάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρησιμοποιούμε τον όρο ενιαίο σύνολο πόρων. Αυτό σημαίνει ότι η μαχημή μονάδα εκπαιδεύεται και διατηρείται και για εθνική χρήση. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εκπαίδευση και άσκηση σε πολυεθνικό περιβάλλον προσθέτει αξία. Αλλά πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι οποιασδήποτε μάχημη τακτική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εθνικούς σκοπούς. Ε, οπότε πρέπει να ε, διατηρείται ασκημένη, πρέπει να διατηρεί τι ασκήσει τη. Ευχαριστώ. Gentlemen, use your earphones, please. speak Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ, θα μιλήσω στα τσέχικα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Σας ευχαριστώ γιατί μίλησατε πολύ ανοιχτά μαζί μας και μας εμπνέει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για την προετοιμασία αυτού του κομματιού της συνεδριασής μας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ όλες και όλους που συμμετείχατε στη συνεδρίαση αυτή. Δεν κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης, γιατί έχουμε και αύριο συνεδρίαση. Απλά διακόπτουμε. Για απόψε. Καλό βράδυ.